Ο Πρόεδρος, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. στη σημερινή μας συνεδρίαση. Σχόλια επί της ημερησίας διατάξεως. Όχι. Δεύτερο. Δύο ανακοινώσεις. Πρώτη. Του χρόνου οι συνεδριάσεις μας θα είναι διαφορετικά χρονικά τοποθετημένες θα είναι πιο συνδεδεμένες οι ημερομηνίες. Γιατί έχουμε μισή μέρα σήμερα, είχαμε μισή, μισή μέρα πριν από λίγες μέρες. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Δεν ξέρω κατά πόσον έχουν καταλάβει τις ημερομηνίε οι άλλες ε, επιτροπές, αλλά νομίζω ότι για όλους μας είναι προτιμότερο να μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, να, είμαστε, να, δραστηριοποιούμε, να δραστηριοποιούμε θα πούμε στις εκλογικές μας περιφέρειες, παρά να ερχόμαστε οπωσδήποτε εδώ για μισή μέρα μόνο συνεδρίαση. Έχουμε τώρα το ξεκάθαρη πλέον εικόνα για τα εκλογικά αποτελέσματα στην Αίγυπτο και παρά τις επανειλημμένες καταμετρήσεις ο Μπεν Μάουζι παίρνει την πλειοψηφία Το χρονικό αυτό διάστημα ωστόσο εκμεταλλεύτηκε ο στρατό ώστε να περικόψει τι αρμοδιότητε του Προέδρου. Πρέπει να δούμε τώρα εάν όντω θα συμφωνήσουν ή θα υπάρξουν πάλι ρήγματα μέσα στην ίδια την Αιγυπτιακή κοινωνία. Πάντως με ικανοποιεί η δήλωση του Πρόεδρου Μορουζή που είπε ότι είναι πρόεδρος όλων των Αιγυπτίων, αυτό με καθησυχάζει για τους χριστιανούς. είναι σημαντικό να διασφαλίζονται τα δικαιώματα όλων των πολιτών και να μην υπάρξουν ρήξεις μέσα στην Αιγυπτικιακή κοινωνία που να οδηγήσουν σε ενδεχομένως πολύ δυσάρεστες εξελίξεις. Σχόλια δικά σας επ' Όχι. Ακολουθούν Ακολουθεί το θέμα της Κούβας. Συνεχιζόμενη καταπίεση από πλευράς του καθεστώτος κατά των λευκών κυριών, στην Πλάνκο. Ο κύριος Καμίνσκι είναι παρόν. Παρακαλείται να κάνει μια σύντομη εισαγωγή στην, στην γραπτή αυτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι στα αγγλικά, ο Σκεμίνσκι, Καμίνσκι, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να θέσω ένα θέμα που αγγίζει την καρδιά των ε, δικαιωμάτων, ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα. Η γραπτή μου ερώτηση προς την κυρία Κάθριν Άστον αναφέρεται στη συγκεκριμένη περίπτωση το, τον, της καταπίεσης σε βάρος των ε, λευκών κυριών που αυτές οι γενναίες γυναίκες συνεχίζουν να αγωνίζονται για τα δικαιώματα και την απόλυση των ε, ανδρών, γαμπρών, πατεράδων τους κλπ. Πολλές από αυτές έχουν ε, ρηχθεί στις φυλακές, έχουν υποστεί κακομεταχείριση και τα σπίτια τους έχουν ερευνηθεί και καταστραφεί από τους ανθρώπους του Κάστρο. Ας δούμε τα γεγονότα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κούβας, ένα τρίτο όλου του εμπορίου και το μισό περίπου των άμεσων αλλοδαπών επενδύσεων. Πάνω από του μισού τουρίστε που πάνε στην Κούβα προέρχονται από την Ευρώπη. Αυτά θα έπρεπε να σημαίνουν καταρχήν ότι για την Κούβα, για την Αβάνα δηλαδή, η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη μια ένωση δημοκρατικών κρατών όπως εμείς να θεωρούμε ότι η ελευθερία είναι η πρώτη στην προτεραιότητα. Παρόλο που λέμε ότι ένα κατά προτεραιότητα στόχων για τι εξωτερικέ δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ενίσχυση των δημοκρατικών συστημάτων και η υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, παρόλα αυτά η παράληψη να αναλάβουμε δράση δείχνει ότι στην ουσία μα αρκεί το business as usual με την Κούβα. Υπερβολικά συχνά μα τυφλώνει η ομορφιά του εξωτικού αυτού νησιού και δεν βλέπουμε τι γίνεται, τι σημαίνει ζωή στην Κούβα. Φτώχεια, φόβος και κρατική τρομοκρατία. Από την Μαύρη Άνοιξη του 2003 πολλές μανάδες πέθαναν χωρίς να δουν να απολύονται τις φυλακές ή γη τους. Οι οικογένειες καταστρέφονται, παιδιά μεγαλώνουν χωρίς ε, πατεράδες και γυναίκες χωρίς συζύγους. Το 2009 το Συμβούλιο επανέλαβε την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει έναν διάλογο βασισμένο σε μια προσπάθεια να επιτευχθούν αποτελέσματα. Ρωτώ, πού είναι αυτά τα αποτελέσματα. Δυστυχώς δεν προσαρμόζουμε τις πολιτικές μας στα γεγονότα που συμβαίνουν επί τόπου. Πάνω από 40.000 συλλήψεις αναφέρθηκαν για το 2011 με το πολύ 1800 στην προηγούμενη χρονιά έχει έρθει η ώρα που οι Κουβανοί θέλουν να αναλάβουν την, την διεύθυνση των, ε, ε, της πατρίδας τους. Ο Κάστρο είχε πει κάποτε ότι θα, η ιστορία θα μου δώσει άφεση. Όχι, η ιστορία δεν θα σου δώσει άφεση. Θα σε καταδικάσει ως δολοφόνο, ως εγκληματία που καταπάτησε τα ανθρώπινα δικαιώματα του κουβανικού λαού για πάνω από μισό αιώνα. Εγώ ωστόσο πιστεύω ότι η ιστορική εκείνη μέρα έρχεται, φτάνει, όταν οι Κουβανοί θα ανακτήσουν την ελευθερία τους και τότε ο Κάστρο θα δικαστεί. Και μετά από αυτή την ημέρα της κρίσης θα μας ρωτήσουν τι κάνατε εσείς όταν μας πετούσαν στις φυλακές. Μας ανάγκασαν να, σιγά, σιγήσουμε και μας εξόρισαν. Πού βρισκόσασταν εσείς οι Ευρωπαίοι όταν μας στέρισαν την αξιοπρέπειά μας. Και είμαι βέβαιος ότι οι λευκές κυρίες θα ρωτήσουν τι κάνατε εσείς Ευρωπαίοι όταν οι αδελφοί μας, οι πατεράδες μας, οι σύζυγοί μας ρίχνονταν στις φυλακές του Κάστρο. Για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει περισσότερη υποστήριξη και αλληλεγγύη με τους ε, κουβανούς αντιφρονούντες και με τους οικείους τους. Σε προσωπική βάση το μόνο που μπορώ να πράξω είναι να απευθυνθώ στο εγκληματικό καθεστώ του Κάστρο και να του πω τα λόγια εκείνα του Αβραμ Λίνκολν. Όσοι στερούν την ελευθερία των άλλων δεν την αξίζουν οι ίδιοι. Συμπεραίνοντα, πιστεύω τα λόγια εκείνα που είχαν ακουστεί στην κομμουνιστική Πολωνία του 1979 από, τότε, από τον Ιωάννη Παύλο τον δεύτερο, τον μεγαλύτερο των συμπατριωτών μου, που είχε πει «Ας έλθει εδώ το πνεύμα και ας αλλάξει το πρόσωπο της χώρας αυτής». Κάτι το οποίο έγινε λίγο μετά. Ελπίζω ότι τα ίδια αυτά λόγια και το ίδιο αυτό πνεύμα θα πνεύσει και στην Κούβα και θα αλλάξει την εικόνα της χώρας αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και σας κύριε συνάδελφε. Παρακαλώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλλον συγγνώμη. Ε, παρακαλώ την ε, εξωτερική υπηρεσία. Την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων να λάβει το λόγο. Βρισκόμαστε εδώ σε μια διαδικασία όπου εάν δεν απαντήσει μέσα σε μια τακτή προθεσμία η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων, ο ερωτών μπορεί να φέρει το θέμα ενώπιον τη Επιτροπή Εξωτερικών. Αυτό έχει συμβεί τώρα. Αυτό αποτελεί και μια υπόδειξη βέβαια προ την Επιτροπή Εξωτερικών Δράσεων να απαντά εντό των προθεσμιών στι ερωτήσει. Έχετε τώρα την ευκαιρία να τοποθετηθείτε. Ναι, η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στην απάντηση που έλαβε ο αξιότιμος βουλευτής την 21η Μαΐου και η οποία πραγματευόταν ακριβώς το θέμα που αποτελεί αντικείμενο της προφορικής του ερώτησης, της εγγραφής του συγγνώμη ερώτησης. Η παρέμβαση του αξιότιμου βουλευτή σήμερα βέβαια ήταν λίγο ευρύτερη. Δηλαδή αναφέρθηκε σε θέματα τα οποία δεν περιείχε η γραπτή του ερώτηση. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν κύριε Πρόεδρε θα δώσω το λόγο στον κύριο Καλογύρου, ο οποίος είναι ο ατματάρχη ε, για την, ε, υπεύθυνο για την Καραϊβική στην ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και ο οποίος μπορεί να απαντήσει ενδελεχέστερα στην ερώτηση του κύριου Βουλευτού. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα απλά να επαναλάβω ότι το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών κρατουμένων, και της κλιμάκωσης προσωρινών ε, κρατήσεων, ε, συλλήψεων κτλ. Είναι ζητήματα τα οποία γνωρίζει πολύ καλά η υπαρκή εκπρόσωπη και τα παρακολουθεί από κοντά. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι θεμελιώδει ελευθερίε είναι και στην καρδιά των σχέσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτε χώρε, μεταξύ αυτών βέβαια και με την Κούβα. Από το 2008 και μετά έχουμε πολιτικό διάλογο με την Κούβα και έχουμε χρησιμοποιήσει κάθε δυνατή ευκαιρία για να θέσουμε στο πλαίσιο αυτό του διαλόγου τα ζητήματα αυτά προς τις ε, αρχές της Κούβας. Αλλά το έχουμε πράξει και σε άλλα επίπεδα, δηλαδή στο επίπεδο της αντιπροσωπείας μας ε, στην Αβάνα, σε επαφές που έχουμε με τις ε, κουβανικές αρχές. Επίση, η αντιπροσωπεία μα, η αποστολή μα στην Αβάνα παρακολουθεί πολύ προσεκτικά όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι σε επαφή με τις ομάδες ε, όλες ε, που συμμετέχουν, όπως και βέβαια και με τις ε, ντάμας ντεμπλάνκο της κυρίας τα Λευκά. Δεν μπορεί κανείς να λάβει να πιστωθεί μάλλον μεμονωμένα την αλλαγή κατάστασης στην Κούβα ο διάλογος, ο πολιτικός, κατόπιν επιμονής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα των πολιτικών κρατουμένων, σε κάποιο βαθμό έφερε κάποια αποτελέσματα και μάλλον έχει και συμβάλει στην απελευθέρωση της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτικών κρατουμένων. Ολοκληρώνοντας να πω απλά, όπως και ξεκίνησα, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα παραμένουν στην καρδιά, στο επίκεντρο των σχέσεων με όλο τον κόσμο με όλες τις χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένες και της Κούβας. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ κυρία Γκόμες. Στα αγγλικά. Θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να ερωτήσω την Κομισιόν. Συγγνώμη, την εξωτερική υπηρεσία. Αν μπορεί να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το είδος επαφών που διατηρεί η αντιπροσωπεία, Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία στην Κούβα με τις οργανώσεις αυτές αντιφρονούντων συμπεριλαμβανομένων των λευκών κυριών. Και επανέρχομαι σε κάτι που είπε ο Καμίνσκι πριν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται εκεί και τάσεται υπέρ των αντιφρονούντων Μάλιστα το κοινοβούλιο έχει, έχει χορηγήσει το βραβείο Ζαχάροφ στη Ντάμαστε Μπλάνκο για να ενισχύσει τη φωνή τους. Και γνωρίζουμε ότι υπάρχει βέβαια διαφορά ύφου μεταξύ κοινοβουλίου και άλλων θεσμικών οργάνων, αλλά το κοινοβούλιο δικαίω έθεσε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το έχει λάβει βέβαια πολύ σοβαρά υπόψη, και την υποστήριξη προσφέρει σε κουβανούς ακτιβιστές και ακτιβίστες ιδίω τη Ντάμα Τεμπλανκό. Η ερώτησή μου είναι, από πλευρά αντιπροσωπεία στην Κούβα, όχι μόνο οι επαφές με τις αρχές. Δέχομαι ότι όντως οι επαφές αυτές ίσως να έχουν οδηγήσει στην απόλυση ορισμένων από τους πολιτικούς κρατουμένου. Αλλά τι είδους υποστήριξη δίνουμε σε αυτές τις οργανώσεις στην Κούβα. Στην πρόσφατη συνάντηση με τους Αμερικανούς συναδέλφους μας στην ε, Κοπενχάγη, μεταξύ των οποίων υπάρχει και μια πολύ ισχυρή φωνή υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Κούβα, του Ντία Μπαλάρτ, είχα την ευκαιρία να ανταλλάξω απόψεις μαζί του και αντελήφθη ότι αλλάζει η κατάσταση. Το δέχεται και ο ίδιος ότι δηλαδή η πολιτική αποκλεισμού, το εμπάργκο, δεν έχει αποδώσει και το αντίθετο μάλιστα. Αλλά λόγω των αλλαγών που εξελίσσονται, που υπάρχουν και γίνονται στην Κούβα, και όλοι περιμένουν πότε θα πιθάνει ο Φίντελ Κάστρο, αλλάζει η διάθεση του κόσμου και ευκαιρίες θα υπάρχουν για αυτούς που αγωνίζονται υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Είναι λοιπόν σημαντικό το Κοινοβούλιο να παραμείνει σε πρωτοπόρο θέση και η υπηρεσία εξωτερικών δράσεων να παραμείνει σε επαφή με τους ακτιβιστές στην Κούβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να θυμίσω στα μέλη της Επιτροπής ότι η Κούβα είναι μοναδική χώρα της Λατινικής Αμερικής που δεν δεσμεύεται με καμία συμφωνία συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η ανομαλία δεν οφείλεται, κατά την ταπεινή μου γνώμη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν η ερώτηση του κυρίου Καμίνσκι ε, επικαλείται τη συνείδηση όλων μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπροστά σε μία κατάσταση παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως είναι αυτό των θεμελιωδών δικαιωμάτων του θεμελιώδου δικαιώματος του να μπαίνει και να βγαίνει κάποιος ελεύθερα στη χώρα του δεν μπορεί να τύχει ούτε αμφίσιμης απάντησης ούτε γραφειοκρατικής απάντησης. Εμείς πρέπει να είμαστε συνεπείς με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο έχει, δώσει, έχει αποδώσει τρεις φορές το βραβείο Ζαχάροφ στην αντιπολίτευση της Κούβας στον Κιγέρμο Φαρίνια, στις γυναίκες με τα άσπρα και σε κάποιον άλλον, ο κανένας από τους τρεις δεν ήρθε να το πάρει. Εγώ ήμουνα ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας συνεργασίας με την Κεντρική Αμερική και την Κούβα. Εγώ πάντα ήθελα να έχουμε διάλογο με τις αρχές και με το λαό της Κούβας. Αλλά κύριε πρόεδρε, ε, είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό όταν έχουμε... Όταν θέλουμε να θεσπίσουμε έναν επικοδομητικό διάλογο με την Κούβα, να υπάρχει μια αναγνώριση των αρχών του Κοινοβουλίου, να μπορούν όσοι είναι δικιούχοι αυτού του βραβείου να έρχονται εδώ και να το παραλαμβάνουν. Το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μάλιστα όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ορίσει έναν ειδικό αντιπρόσωπο ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν, ε, αυτά τα δικαιώματα δεν θα πρέπει να τα δούμε μόνο σε σχέση με μια χώρα αλλά παγκοσμίω. Ε, εμείς ε, ε, ενδιαφερθήκαμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κατάσταση κράτησης των κουβανών στις Ηνωμένε Πολιτείες. Εμείς όμως πρέπει να διεκδικήσουμε και το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα του να μπαινοβγαίνει κανείς δηλαδή ελεύθερα από τη χώρα του και στη χώρα του και να μπορέσει το κοινοβούλιο κάποτε να δώσει και το βραβείο, να αποδώσει πλέον το βραβείο στους ενδιαφερόμενους. Πολλοί από εμά ε, θέλουμε να εξομαλύνουμε τις, τις σχέσεις μας, αλλά και οι κουβανικές αρχές ε, πρέπει να, δώσουν, να κάνουν και αυτές ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και να επιτρέψουν την έξοδο από τη χώρα σε αυτούς που πρέπει να τους δοθεί το βραβείο. Ε, ξέρω ότι πρέπει να αλλάξει η κοινή θέση του Συμβουλίου για αυτό το θέμα. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να δοθεί η άδεια στους βραβευμένους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κυκλοφορούν ελεύθερα. Τώρα τα υπόλοιπα για την εξέλιξη της Κούβας, αν θα ακολουθήσει ένα μοντέλο κινέζικο ή βιετναμικό ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι είχαμε κάποια πρόοδο, αποφυλακίστηκαν άνθρωποι οι οποίοι ποτέ δεν θα έπρεπε να είχαν φυλακιστεί αλλά επιμένω. Όλοι αυτοί οι οποίοι βραβεύτηκαν για τον αγώνα τους να μπορέσουν να έρθουν στο κοινοβούλιο και να παραλάβουν το βραβείο τους. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση πρώτα σχετικά με την επισήμανση του κ. Σαλαφράνκα. να κάνουμε την προσπάθεια είτε εδώ είτε στην Κούβα να κάνουμε την απονομή του βραβείου. Έχω απορρίψει ή έχουμε απορρίψει και θα απορρίψω κάθε πρόσκληση από πλευρά Κάστρο ε, στην Κούβα εάν δεν έχουμε τη δυνατότητα να απονείμουμε προσωπικά το βραβείο στους βραβευομένους. Παρόμοια η περίπτωση με τους βραβευθέντες από τη Βιρμανία. Μπορεί και το Προεδρείο του Κοινοβουλίου να επανεξετάσει ποιοι βραβευθέντες δεν μπόρεσαν να παραλάβουν τα βραβεία τους και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και ίσως μπορεί να μας βοηθήσει και η Επιτροπή, ε, Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων. Και να δούμε και την επίσημη απάντηση της Λέδης Άστον που λέει ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν επαναλάβει σε διάφορες περιπτώσεις την ανάγκη η Κούβα να σεβαστεί τα δικαιώματα του κουβανικού λαού. Μπορείτε να μας πείτε πού έγκυται η πρόοδος περί της οποίας μιλούν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τις επαφές και τις ε, δράσεις που αναλαμβάνουμε σε σχέση με την ειρηνική αντιπολίτευση της Κούβας, μπορώ να σας πω ότι η αντιπροσωπεία διατηρεί έναν δραστήριο διάλογο, δηλαδή έρχονται άνθρωποι στην αντιπροσωπεία μας και μιλούν με την αντιπροσωπεία μας, μας μεταφέρουν μηνύματα μέσω αυτού του διάβλου, ενώ επίσης και μέλη της αντιπροσωπείας συναντούν και συνομιλούν ε, με μέλη της ελληνικής, της ελληνικής αντιπολίτευσης. Επίσης και με τις άλλες πρεσβείες ε, στην Αβάνα, η αντιπροσωπεία ε, συμμετέχει και αυτή στην ομάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία όχι μόνο διατηρεί επαφέ με το κίνημα των αντιφρονούντων, αλλά καλεί τακτικά και άνθρωπου στις συναντήσεις της, στις συνεδριάσεις της. για να συζητά διάφορα ζητήματα μαζί τους. Τώρα, τι συγκεκριμένε ενέργειε αναλαμβάνουμε για του αντιφρονούντε ή με του αντιφρονούντε. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να εδοθεί στο πλαίσιο ε, της γενικότερης ε, που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι απλά οι υπηρεσίες δράσεις δράσης ενέργειες ε, που γίνονται με την κοινωνία των πολιτών. Υπάρχουν διάφοροι φορεί, διάφορε οντότητε και τα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν διαφόρους διάβλους και μέσα που μπορεί να είναι ή να μην είναι προσαρμοσμένα για την επίτευξη αποτελεσμάτων, γιατί πρέπει να έχουμε κατά νου πάντοτε και την ε, ασφάλεια και την προστασία των προσώπων. Μα τέτοιο το ερώτημα αν υπάρχει κάποια συμφωνία με την Κούβα. Όχι, πράγματι δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Είναι μια από τι ελάχιστε χώρε στον κόσμο με την οποία δεν έχουμε καμία συμφωνία. relations with Cuba. Σήμερα οι σχέσεις μας με την Κούβα βασίζονται στην κοινή θέση. Υπάρχει μια συζήτηση για το κατά πόσο η κοινή θέση πρέπει να παραμείνει ως έχει ή να αντικατασταθεί από συμφωνία σε κάποια χρονική στιγμή. Αυτή η συζήτηση συνεχίζεται εδώ και καιρό στο επίπεδο του Συμβουλίου. Είναι διαρρεμένα τα κράτη-μέλη προς αυτό όχι κατά το ίμιση, τα μισά υπέρ, τα μισά κατά, αλλά υπάρχει διάσταση απόψεων. Δεν συμφωνούν όλοι. Όλοι πάντως συμφωνούν ότι η γενική στόχη είναι η πραγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπινών δικαιωμάτων στην Κούβα και νομίζω ότι ο στόχος μας και οι θέσεις που λαμβάνουμε είναι με γνώμονα το πώς θα πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η κοινή θέση είναι το καλύτερο εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Μάλλον αυτό πιστεύουν κάποιοι άλλοι. Πιστεύουν ότι διμερεί συμφωνίες με το κατάλληλο περιεχόμενο κάτι που γίνεται με όλες τις συμφωνίες που συνάπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες θα ήταν μια καλύτερη πλατφόρμα για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα με αυτές τις επαφές. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, σχέσεις ε, με το Κοινοβούλιο, πριν από λίγες ημέρες ήμασταν ε, μαζί με τους κουβανούς στη συνεδρίαση της Κεντροαμερικανικής Αντιπροσωπείας και φάνηκε και οι δύο πλευρές να συμφωνούν στο ότι θα πρέπει τα κοινοβούλια να συνομιλούν μεταξύ τους και υπήρξε και πρόταση ενδεχομένως να συμμετάσχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να έχει κάποιο είδους επαφές με το Κουβανικό Κοινοβούλιο. Ο Κουβανός πρέσβης συμφώνησε να μεταφέρει στην Αφάνα το μήνυμα αυτό. Ίσως αυτό θα μπορούσε να είναι και μια δυνατότητα ώστε να απομνημηθεί και το βραβείο Ζαχάροφ ε, στους βραβευθέντες από την Κούβα που δεν έχουν καταφέρει να το λάβουν. Αυτοπροσώπους. Τελευταίο ερώτημα. Μας είπατε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να σημαίνουμε πρόοδο. Εγώ νομίζω ότι η κατάσταση σήμερα πόρο απέχει του να είναι τέλεια, ωστόσο είναι και πολύ διαφορετική σε σχέση με το πώς ήταν πριν από λίγα χρόνια. Μπορεί κανείς βέβαια να συζητήσει το αν είναι πολύ καλύτερη, διαφορετική ή λίγο διαφορετική, αλλά η απελευθέρωση πολιτικοκρατουμέ, κρατουμενου οπως και αν έγινε, από όποιους όρους και αν έγινε, αυτό νομίζω ότι συνιστά κάποιο είδους αλλαγή. Έξω και θα ενθαρρύναμε τις κουβανικές αρχές να συνεχίσουν ε, στο ίδιο αυτό μονοπάτι, να απελευθερώσουν όλους τους πολιτικούς κρατουμένους και να φροντίσουν να γίνονται σεβαστά όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους. Αυτό θα θέλαμε να δούμε στην Κούβα. Ah, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριο Σκαμίνσκι. Ήθελα να πω ότι ικανοποιήθηκα από την απάντηση που έλαβα από το γραφείο της ΥΠΑ ε, της εκπροσώπου. Εκτός από το τελευταίο μήνυμα που έλαβα με αυτό σχετικά με τι επαφέ με αυτό το λεγόμενο κουβανικό κοινοβούλιο. Αγαπητοί φίλοι, δεν υπάρχει κοινοβούλιο στην Κούβα. Υπάρχει ένα διορισμένο όργανο, διορισμένο από το κομμουνιστικό καθεστώ. Αν θέλουμε να μα φέρονται με αξιοπρέπεια ω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ω Κοινοβούλιο τη Ευρώπη που έχει εκλεγεί από του Ευρωπαϊκού Λαού, δεν μπορούμε να δεχθούμε να έχουμε οποιαδήποτε επίσημη επαφή με ένα όργανο το οποίο δεν είναι κοινοβούλιο είναι ένα όργανο διορισμένο από τους δικτάτορες. Κατανοώ ότι πρέπει να εμπλεκόμεθα σε διάλογο με τις κουβανικές αρχές, όπως χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε και τους τρομοκράτες, όπως χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε και τους εγκληματίες που συλλαμβάνουν ομήρους. Τα κατανοώ αυτά. Αλλά μην έρχεστε να μου πείτε ότι οφείλουμε να διατηρούμε επαφές με ένα κοινοβούλιο που δεν αξίζει το όνομά του. Η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω, τελειώνοντας, είναι ότι ανησυχώ πράγματι ότι το θέμα αυτό, το κουβατικό θέμα δηλαδή, μπορεί να αντιμετωπίζεται εδώ στο Κοινοβούλιο ως θέμα αριστεράς ή δεξιάς. Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο. Εγώ παρατηρώ την κατάσταση στην Κούβα πολύ προσεκτικά και γνωρίζω ότι οι κρατούμενοι στην Κούβα προέρχονται από όλα τα ιδεολογικά, από όλους τους ιδεολογικούς χώρους. Φιλελεύθερες φυλακές, στις φυλακές, κομμουνιστές είναι στις φυλακές, αξιοπρέπεις άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερα ε, ορισμένοι από αυτού δεν έχουν καν ιδιαίτερε πολιτικέ πεπιθήσει. Είναι αξιοπρεπεί άνθρωποι και όμω είναι χωμένοι φυλακέ. Εγώ πιστεύω ότι ο αγώνα για την Κούβα είναι αγώνα υπέρ τη πραγματική δημοκρατία. Το λέω διότι έχω πολλές επαφές με κουβανούς αντιφρονούντες. Αυτό που πραγματικά είναι το εκπληκτικό στην περίπτωση αυτή είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν πραγματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πιο πεπισμένοι είναι πεπισμένοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περισσότερο καλύτερη φίλη της Κούβας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μιλώ για ανθρώπους, όπως είπα, από οποιαδήποτε οποιοδήποτε ιδεολογικό πολιτικό υπόβαθρο και είναι τώρα οι άνθρωποι αυτοί χωμένοι στις φυλακές και όμως πιστεύουν στην κοινότητα αξιών μας και εγώ ελπίζω ότι η δική μας κοινότητα αξιών η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει τους κουβανούς να ανακτήσουν την ελευθερία που τους αξίζει. Ωραία. Έληξε εδώ η συζήτηση του θέματος αυτού. Α, ο κύριος και επιθυμεί να αγορεύσει. Όπως ε, είπα και στην προηγούμενη τοποθέτησή μου, εγώ ε, πάντοτε ήμουν πεπισμένος ότι χρειάζεται ε, πάντοτε συζήτηση με την κουβανική κοινωνία και την κουβανική κυβέρνηση. Πρέπει όμως και η, εξωτερική, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να, να βρούμε μία αξιοπρεπή λύση για την απόδοση των βραβείων Ζαχάροφ. Το Κοινοβούλιο είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη, είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει δημοκρατικά το εκτελεστικό όργανο, επικυρώνει σύμφωνα με τη Λισαβόνα τις συμφωνίες συνεργασίας και όπως το είπαμε και στον παλιό, στον πρώην πρεσβευτή της Κούβας, θα πρέπει να βρεθεί μία αξιοπρεπή λύση ούτως ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το είπα και πριν, Τώρα που θα έχουμε και έναν είπα το εκπρόσωπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Κούβα να κάνει αυτή τη χειρονομία και να επιτρέψει στους πολίτες της ε, να βγουν και να ξαναμπούν στη χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα εξετάσουμε ποιοι από τους βραβευθέντες με το βραβείο Ζαχάροφ δεν μπόρεσαν να παραλάβουν το βραβείο τους και μετά θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Εφόσον υπάρχει συμφωνία, οφείλει να συμφωνήσει, ε, οφείλει να εγκρίνει τη συμφωνία δηλαδή, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι στη διακριτική ευχαίρεια του Συμβουλίου η σύναψη και έγκριση της συμφωνίας. Θέλω να έχω λοιπόν ενημέρωση για την εξέλιξη τέτοιων υποθέσεων. δεν μπορεί να συνεχίζεται να ασκείται εξωτερική πολιτική στη βάση μόνο μια κοινή θέση του Συμβουλίου, χωρί να έχει υπάρξει έγκριση και από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, για το θέμα αυτό θα ήθελα να διεξαχθεί γενική συζήτηση. Όπω είπα για το θέμα αυτό, διότι απαιτείται να διευκρινιστεί αν αυτό ισχύει και για άλλες περιπτώσεις, διότι στην περίπτωση αυτή πρόκειται για υπονόμευση των αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου. Έρχομαι στο θέμα υπαριθμών 4, ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στην Λιβύη με τον Αλέξανδρο Κόμιτα Λάμστορφ, που είναι μέλος της ε, ομάδας παρατήρησης των εκλογών στην χώρα αυτή. Βέβαια, αυτά έγιναν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. υπήρχε το Electoral System Project και με συμμετοχή του αναπληρωτή, είχα μάλλον εδώ πρόσφατα τον αναπληρωτή πρόεδρο της Λιβύης, κύριο Αρμπουσόα, και ο Κόμις Λάμστορφ ας μας ενημερώσει Είναι γνωστό άλλωστε γιατί για λόγους τεχνικούς οι εκλογές αναβλήθηκαν για την 7η Ιουλίου. Ναι, ναι, ασφαλώς να σας ενημερώσω, αλλά στα αγγλικά. Και για να κατανοήσουν οι συνάδελφοί μου που βρίσκεται η χώρα τώρα, υπενθυμίζω ότι η πρωτεύουσα Τρίπολη έπεσε στις αρχές του Αυγούστου 2011 και οι εκλογές ήδη προγραμματίστηκαν για τις 7 Ιουλίου, δηλαδή λιγότερο ένα, από ένα χρόνο μετά την πτώση της Τρίπολης. Είναι εξαιρετικά βραχή το χρονικό διάστημα και πιστεύω ότι εξετάζοντας την κατάσταση στη Λιβύη σήμερα οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι παρά τις συνολικές δυσκολίες η πρόοδος της εξελίξεως ήταν καλή σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την εκλογική διαδικασία δεν υπάρχουν σχεδόν συνομιλητές οι οποίοι να θεωρούν ότι απαξιούται η εκλογική διαδικασία και που να μην επιθυμούν να διεξαχθεί ειρηνικά. Η συντριπτική τους πλειοψηφία επιθυμεί να διεξαχθούν ειρηνικά οι εκλογές. Όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, αναβλήθηκε από την 9η Ιουνίου για λόγους όμως και νομικούς και τεχνικούς δεν μπόρεσε να γίνει σεβαστή εκείνη η ημερομηνία της 9ης έκτου δηλαδή. Τώρα όμως υπάρχει αρκετή πεποίθηση ότι θα μπορέσει να γίνει η εκλογή στις 7 Εβδόμου. Για να αλλάξει, να ε, αντικατασταθεί το μεταβατικό κυβερνητικό συμβούλιο από ένα κοινοβουλευτικό όργανο που θα ε, ονομάζεται Γενικό Εθνικό Συνέδριο και αυτό μετά θα διορίσει συνταγματική επιτροπή που θα αποτελείται από 60 μέλη, άνδρες και γυναίκες, που θα συντάξουν ένα πραγματικό σύνταγμα εργασίας για την χώρα. Δηλαδή, λιγότερο από ένα έτος μετά από την πτώση της ε, Τρίπολης και ήδη βρισκόμαστε στα πρόθυρα της ε, συνταγματικής διαδικασίας, δηλαδή στην, ε, στις αρχές της συντάξεως του συντάγματος. Τι έχει γίνει τώρα για να προετοιμαστεί η χώρα από 3,5 εκατομμύρια που δικαιούνται να ψηφίσουν, τα 2,9 έχουν εγγραφεί στους εκλογικού καταλόγους. Πραγματικά σημαντική εξέλιξη. Η προεκλογική εκστρατεία άρχισε στις 18 εκτού, δεν έχει ακόμα ε, αναπτύξει ταχύτητα διότι όλοι όσοι ζούμε εδώ μέσα σε κόμματα γνωρίζουμε πόσο δύσκολες είναι οι προεκλογικές εκστατείες. Όμως τα κόμματα στη Λιβύη άρχισαν να δουλεύουν μοναχά μετά από την επιστροφή των εξορίστων στη Λιβύη, μετά την πτώση δηλαδή της Τρίπολης, δεν υπήρχαν τέτοιες οργανώσεις γιατί ήταν παράνομες υπό το δικτατορικό καθεστώς και χρειάστηκε λοιπόν να τα φτιάξουν από την αρχή όλα, όλες τις υποδομές τους, να νοικιάσουν γραφεία, να αποκτήσουν προσωπικό να αναπτύξουν μια πλατφόρμα προεκλογικής εκστρατείας. Για όλους τους λόγους αυτούς δεν είναι εκπληκτικό λοιπόν που δεν έχει προχωρήσει αρκετά η προεκλογική εκστρατεία και δεν έχει αποκτήσει την ε, απαραίτητη ταχύτητα. Τα κόμματα με τα οποία έχω μιλήσει, 142 είναι συνολικά τα κόμματα, τα πολιτικά κόμματα εκεί, 142 είναι πραγματικά εκπληκτικός ο αριθμός. Ωστόσο, Υπάρχουν ορισμένα κόμματα τα οποία θεωρούνται ότι υπόσχονται περισσότερο σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των εκλογών. Έχω μιλήσει με ορισμένα από αυτά. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι ιδεολογικές τους πλατφόρμες είναι πολύ κοντά, όπως έχουμε αντιληφθεί μέχρι τώρα. Η απόφαση του ψηφοφόρου θα βασιστεί πιθανότατα σε, λιγότερο σε πολιτικές φιλοσοφίες, πολιτικά θέματα, αλλά περισσότερο στο που τοποθετεί το κόμμα απέναντι στον διχασμό σε δυτική και ανατολική της χώρας. Όπως ξέρετε η Βενγάζη ήταν αντίθετη με το καθεστώς του, του Καντάφη περισσότερο και υπάρχει τώρα λοιπόν μια, ε, ένα ρήγμα ανάμεσα στην δυτική και ανατολική ε, ε, Λιβύη. Με ποιο τρόπο κινήθηκαν οι τοπικοί άρχοντες, τι υπόσχονται οι διοικήσεις. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν θα είναι σημαντικότερα από την πολιτική ας πούμε ε, φιλοσοφία ευρωπαϊκού τύπου όπως τη γνωρίζουμε δηλαδή εδώ από τα κόμματα. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση ασφάλειας στην χώρα, εξακολουθεί αυτή να βρίσκεται, να είναι πολύ δύσκολη. Η κεντρική κυβέρνηση δεν ελέγχει ολόκληρη την λιβική επικράτεια. Ξεκολουθούμε να αντιμετωπίζουμε τοπικές πολιτοφυλακές που ελέγχουν την άμεση περιφέρεια επιρροής τους. Αυτό δεν ενοχλεί πάντα τους κατοίκους, διότι αυτές οι τοπικές πολιτοφυλακές εξασφαλίζουν την ε, βασική ασφάλεια, επειδή δεν υπάρχουν άλλες κρατικές ε, δομές. Δεν θεωρείται λοιπόν καταρχήν αρνητική αυτή η εξέλιξη, αντίθετα μάλλον, αλλά μακροπρόθεσμα, όχι σε εκλογικό αλλά σε πολιτικό πλαίσιο, θα είναι σημαντικό οι εθνικές αρχές, θα είναι κρίσιμο μάλιστα, να διασφαλίσουν το μονοπόλιο της εξουσίας. Το κράτος προσπάθησε να το εξασφαλίσει αυτό, δημιουργώντας ε, την λεγόμενη ανώτατη, πολιτική, ε, ανώτατη Επιτροπή Ασφαλείας, που είναι κάπως ενηγματικού χαρακτήρα. Ονομαστικά δηλαδή υποτίθεται ότι έχει 110.000 μέλη, εγώ άκουσα και τον αριθμό 60.000 εγγεγραμμένους στους ε, καταλόγους ε, μισθοδοσίας, αλλά μόνο 5.000 περίπου ε, πάνε πραγματικά να εργαστούν. Η εθνική αστυνομία εξακολουθεί να υπάρχει και λειτουργεί. Η δομή της όμως είναι αδύναμη απέναντι στις βαριά οπλισμένες πολιτοφυλακές και σε ορισμένα τμήματα της ε, Ανώτατης Επιτροπής Ασφάλειας. Ένα θέμα που θα τεθεί είναι η ένταξη στις δυνάμεις αυτές των ε, μαχητών. Αν αυτό θα καταστεί δυνατόν, θα εξαρτηθεί από τις οικονομικές πρόπτικες της χώρας. Της χώρας. Λόγω των υψηλών ε, εσόδων από το πετρέλαιο, το καθεστώς Καντάφη έδινε αυτονα παροχές. Ε, οι άνθρωποι είχαν τέσσερις και πέντε δουλειές που δεν πήγαιναν σε όλες βέβαια, εισέπραταν όμως από όλες. Και οι αλλαγέ αυτέ τώρα είναι σημαντικέ βέβαια προκλήσει για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Ασφαλώ τα έσοδα από το πετρέλαιο θα συνεχίσουν να υπάρχουν με ένα πληθυσμό όμω που είναι κατά 40% λιγότερο των 18 χρονών. Ασφαλώ αντιλαμβάνεται κανεί ότι η δημιουργία θέσεων εργασία και οικονομική προοπτική είναι ζήτημα και μεταξύ άλλων και αξιοπρέπεια και αυτοσεβασμού τη χώρα. Τώρα υπάρχουν Πηγέ που ενδέχεται, από όπου ενδέχεται να προκύψουν δυσκολίε για τι εκλογέ. Οι περισσότεροι συνομιλητές μου δεν αναμένουν ή οδήποτε αποσταθεροποίηση σε εθνική κλίμακα. Υπάρχουν ωστόσο θύλακοι δυσαρέσκειας, ας το πω έτσι. Υπάρχει ένα πολύ... Υπάρχει ένα τμήμα ε, ε, ομοσπονδιόφιλων, να το πω έτσι, φεντεραλιστών, οι οποίοι έχουν ε, ε, προκαλέσει, έχουν ε, κατέλθει σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στη Βενγκάζη κλπ. Υπάρχουν κάπου κάπου και εκδηλώσεις αλαφιστών, πάλι κυρίως στα ανατολικά της χώρας, γύρω από την Τέρνα, Ε, έκαναν ε, εκδηλώσεις επίσης ε, αποδοκιμασιών και στην Βενγάζη. Πάντως, κανένα από τα κινήματα αυτά δεν θεωρείται αρκετά ισχυρό είτε αρκετά πολυάριθμο για να μπορέσει να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση. Όλα αυτά που είπα είναι βέβαια προκαταρκτικές εκτιμήσεις. Οι εκλογές αναπτύσσουν ίδια δυναμική από το 1965 δεν, έχει, δεν έχουν γίνει εκλογέ ε, στη Λιβύη. Θα δούμε λοιπόν πώ θα πάνε τα πράγματα. Θα ολοκληρώσω λέγοντα δύο ακόμη πράγματα. Πρόκειται για ένα ε, λαό που θέλει ε, να επιτύχουν οι εκλογέ. Έχουν ήδη γίνει δύο τοπικέ, Βενγκάζη και Μισράτα. Αλλά και η ορολογία της δημοκρατίας δεν είναι γνωστή στον, σε πολλούς ε, Λίβιου όταν μιλεί κανεί για κοινοβούλια, κόμματα κτλ. Αυτά είναι πράγματα που ακούν πρώτη φορά. Πρόκειται λοιπόν για μια απαρχή μια διαδικασία και όχι για το τέλο με τι εκλογέ αυτέ. Και το άλλο που είναι περισσότερο εσωτερική κατανάλωση δική μα, όπως θα είδετε είμαι επικεφαλή ομάδας παρακολούθηση παρατήρηση των εκλογών. Θεωρήσαμε ότι για λόγους ασφαλείας δεν θα στέλναμε μια ομάδα παρατήρηση εκλογών που να καλύπτει όλη την επικρατεία. Την επικρατεία πρόκειται περισσότερο λοιπόν για assessment mission, αξιολόγηση των εκλογών. Και αυτό είναι κάτι το νέο, γιατί ε, ε αυτή τη ομάδα ηγείται ευρωβουλευτή, εγώ δηλαδή εν προκειμένου, και είναι κάτι διαφορετικό από τι συνήθει αποστολέ παρατήρηση εκλογών και τη αξιολόγηση, βέβαια που συνήθω είναι πολύ μικρότερε, αλλά λόγω τη εγκύτητα και τη σημασία τη χώρα αποφασίστηκε να ε, κάνουμε αυτό για να δώσουμε επαρκή ορατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτόπου και να δείξουμε ότι θέλουμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους Λίβιους στην πορεία τους αυτή. Αυτές είναι οι πρώτες μου λοιπόν προκαταρκτικές επαναλαμβάνω παρατηρήσεις για το θέμα κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γκόμης. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αλεξάνδρ Λάμστορφ για την πολύ καλή αυτή ενημέρωση. όλα όσα είπε συμπίπτουν απόλυτα και με το πώς εγώ έχω ε, αντιληφθεί την όλη κατάσταση, ε, όχι για τις εκλογές που αποτελεί δική του αρμοδέτα, αλλά σε ό,τι την ευρύτερη εικόνα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι περί αυτού ακριβώς πρόκειται. Δηλαδή όλοι κατανοούμε ότι οι εκλογές αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές υπό την έννοια ότι θα επιτρέψουν ε, σχηματισμό ενός ε, σώματος που συνέχει, στη συνέχεια θα ξεκινήσει εργασία για τη σύνταξη συντάγματος. Και θα πρέπει βέβαια να ε, προκύψει και από τις εκλογές μια κυβέρνηση η οποία θα έχει την νομιμοποίηση που μόνο εκλογές μπορούν να δώσουν. Σε ό,τι αφορά τώρα το ενδεχόμενο μποϊκοταρίσματος ε, των ε, εκλογών, ε, νομίζω ότι όλοι θα αντιληφθούν ότι είναι πολύ σημαντικές για το μέλλον της χώρας και δεν θα κάνουν κάτι τέτοιο. Ανέφερε μια μικρή ομάδα ο Αλεξάνδερ, οι οποίοι ζητούν ομοσπονδοποίηση. Ο κύριος Αχμέντα Ζανούση, που έχει βραβευτεί πέρυσι, βραβεύτηκε με το βραβείο Ζαχαροφίνο επικεφαλής Στη Βενγκάζη είχαμε κάποιες συναντήσεις ε, και με άλλους δέκα. Ξέρουμε ποια είναι, ποιες είναι οι επιδιώξεις τους. Και στη Βενγκάζη ακόμη και κάποιοι οποίοι λένε στεναρά ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί η Βενγκάζη και να ε, γίνουν επενδύσεις γιατί είχε παραμεληθεί πολύ επί εποχής Καντάφη. Ακόμη και αυτοί θεωρούν ότι είναι εντελώ περιθωριακή ομάδα του Αλζανούση, δηλαδή δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις ε, των κατοίκων της Βενγκάζη. Πρέπει να σας πω ότι στι συναντήσει που είχα μαζί τους, σχεδόν ε, μας ζήτησαν συγγνώμη Μας είπαν ε, ότι υπάρχει πράγματι και ένα Ισλαμικό αντίβαρο, έχουμε τους αλαφιστές οι οποίοι οργανώνονται, η μουσουλμανικοί αδελφότητα επίσης, ε, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αιγύπτου, αλλά όχι με τρόπο που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα το πρόσχημα για τη δημιουργία ενός ε, αντικινήματος. Παραλαμβάνω κατά την άποψή μου ούτε και οι κάτοικοι της Βεγγάζης είναι υπέρ αυτής της ε, Άρα νομίζω ότι δεν τίθεται ζήτημα διαίρεσης ε, Δύσης Ανατολής. Τώρα, να μιλήσω συνολικά για το θέμα της ασφάλειας. Όπως είπε ο Αλεξάνδερ, υπάρχουν πολλά προβλήματα στον τομέα αυτό, δεν είναι καθόλου καλή κατάσταση, διότι όπως είπε η κεντρική κυβέρνηση δεν ελέγχει τόσο όλοι τις επικράτες. Ουδής όμως ε, το ελέγχει. Πρώτα απ' όλα, διότι το μεγαλύτερο μέρος της επικράτησης είναι έρημος και εκεί που κατοικούν άνθρωποι, στα μεγάλα κέντρα, υπάρχει ηρεμία, αλλά υπάρχουν θύλακοι. Πράγματι υπάρχουν αυτές οι, πολιτικές, οι πολιτοφυλακές, οι παραστρατιωτικές ομάδες που συγκροτήθηκαν για να ανατρέψουν την κυβέρνηση, αλλά τώρα έχουν διατηρήσει τον οπλισμό τους, ε, ε, δεν έχουμε βέβαια ε, κάποιες εξεγέρσεις με κεντρική διοίκηση όπως είχαμε στο Αφγανιστάν για παράδειγμα. Είναι πιο πολύ μεμονωμένα αυθόρμητα περιστατικά. Ακούσαμε ε, και πρόσφατα ε, να γίνονται κάποιες μάχες μεταξύ κάποιων φυλών, αλλά είναι πάρα πολύ ε, εντοπισμένες, ε, περιορισμένες σε ένα συγκεκριμένο τόπο διαμάχες μεταξύ φυλών. Άρα έρχομαι στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά και τώρα και στο μέλλον αν ενισχύσει την εθνική συμφιλιωτική προσπάθεια για να σταματήσουν αυτές οι φιλετικές αντιμαχίες και αντιπαραθέσεις. Αυτό το είδα και την τελευταία φορά που πήγα εκεί. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα ε, διότι συνάντησα και είδα ε, πράγματα μεταξύ τους ε, κατοίκους της Μιζάτα και της ε, Τάουρκ. Υπάρχουν μακρά, υπάρχει μια μακρά ιστορία αντιπαλότητας μεταξύ αυτών των δύο πόλεων. Η πόλη αυτή όμως σχεδόν έχει καταστραφεί ολοσχερός πια και οι κάτοικοί της περιφέρονται από εδώ και από εκεί. Είναι μια τραγική, ίσως η πιο τραγική κατάσταση που βίωσα εγώ εκεί. Και κάτι και των δύο πόλεων ε, είναι θύματα αποτρόπαιων εγκλημάτων, βιασμοί, ε, κατηγορούνται οι κάτοικοι της ΤΑΟΡΚ ότι βίασαν άντρες και γυναίκες στη Μισράτα. Πρέπει να υποδοθεί δικαιοσύνη. Και στον τομέα αυτό Πραγματικά νομίζω ότι και εμείς μπορούμε να κάνουμε πολλά και να βοηθήσουμε τους ε, Λίβιους για να προβούν στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και του δικαστικού συστήματος. Ίσως θα πρέπει να δούμε και με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τι μπορούμε να κάνουμε. Τέλος, θα ήθελα να πω το εξής. Έχω την εντύπωση ότι ευτυχώς, ευτυχώς πια έχουμε έναν πρέσβη από το Μάιο και με ικανοποιεί ιδιαίτερα μέχρι τώρα δουλειά που κάνει εκεί. Βέβαια υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερο συντονισμό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να στελεχωθεί η υπηρεσία. Δεν υπάρχει ακόμη επαρκέ προσωπικό. Δεύτερον, επαναλαμβάνω, καλύτερο συντονισμό και εδώ στι Βρυξέλλε και δι' μεταξύ υπηρεσία εξωτερική δράση και κομισιών. Πρέπει να κινητοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κάνει τη δουλειά που ξέρει να κάνει. Και υπάρχουν και απαραίτητοι πόροι γι' αυτό. Και επαναλαμβάνω, συντονισμό. και με τα κράτη-μέλη. Έχω διανύμει μία έκθεση στους ενδιαφερόμενους συναδέλφους όπου αναφέρω τα πορίσματα της τελευταίας μου επίσκεψης στη χώρα. Και ουσιαστικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης θέλουμε να κάνει τη δουλειά της, να συντονίσει τα κράτη-μέλη δηλαδή. Τα κράτη-μέλη ουσιαστικά ξανακάνουν τα ίδια ό,τι έκαναν και στο παρελθόν. Δηλαδή, η Γαλλία προσπαθεί να, προσπαθούσε να πουλήσει στο Καντάφι ένα πυρηνικό εργοστάσιο, η Ιταλία με τον Περλουσκόνη ήταν, είχαν ψύχος με το θέμα της μετανάστευσης. Και τελικά προσπαθούμε να φτιάξουμε μια συμφωνία πλαίσιο. Και βλέπω ότι επανέρχονται στα ίδια. Οι λιβικές αρχές από ό,τι είδα γύρισαν και είπαν, μα τι είναι αυτό η ασφάλεια των συνόρων. δεν μπορείτε εσείς οι Ευρωπαίοι αντί να έχετε τρεις-τέσσερις προτάσεις, προερχόμενες δηλαδή από κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχετε μόνο μία. Αυτό χρειαζόμαστε πράγματι. Και πρέπει να παρακαλέσουμε την Λέδια Άστον να μην τρέπεται και να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να συντονίσει καλύτερα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Λάμστορφ όχι μόνο για τις πληροφορίες που μας έδωσε σχετικά με τις εκλογές στη Λιβύη αλλά για το ότι θέλησε να είναι και επικεφαλής αυτής της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για να σηκώσει και το προφίλ της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πήγε να παρακολουθήσει όλη αυτή τη διαδικασία εκδημοκρατισμού σε αυτή τη χώρα. Είναι φανερό ότι γνωρίζουμε και από τις επισκέψεις διαφόρων στελεχών της Λιβύης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γνωρίζουμε λοιπόν την κατάσταση στη χώρα και καταλαβαίνουμε ότι η οργάνωση μιας εκλογικής ε, διαδικασίας μέσα σε αυτή την περίοδο θεσμικής ε, ε, ε μεταπολίτευσης δημιουργεί πρόβλημα. Δεν είναι εύκολο να γίνει. Θα ήθελα να ξέρω όμως αν έχει στοιχεία για το ποια μέσα θα κινητοποιήσει ο ΙΕ, αν θα υπάρξουν άλλοι παρατηρητές από την Αφρικανική Ένωση, από την ε, Ισλαμική Συνεργασία, από άλλους διεθνείς οργανισμούς, ε, τι ρόλο θα παίξουν τα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίσης, πώς θα χρηματοδοτηθούν τα πολιτικά κόμματα πάνω από 50, όπως είπε ο κύριος Λάμστορφ. Είπε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αλεξάνδρ για την ενημέρωση και συμφωνώ, ήταν εντυπωσιακή ενημέρωση ε, και για την επισκέψη του ε, αντιπρόεδρου της Εγώ βέβαια έχω κάποιες δικές μου απόψεις ε, μετά την απαγωγή συγγνώμη, κάποιων εκπροσώπων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, η Σαρία επίσης ε, που θα μπει στο Σύνταγμα και σίγουρα θα εμπνεύσει και η νίκη του Μόρση στην Αίγυπτο. μεταβατική δικαιοσύνη, πάρα πολλά θέματα. Ε, πώς θα αποταθεί δικαιοσύνη για όλα αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα της εποχής ε, Καντάφη, πώς θα μπορέσουν να συμφιλειωθούν ε, οι πόλεις, ε, οι φατρίες, οι φυλές κτλ. Και το τεράστιο ζήτημα ασφάλειας στο Νότο βέβαια ε, από το Κατάρ και τις χώρες του κόλπου μπήκαν τεράστιες ποσότητες όπλων που τώρα είναι στα χέρια των Τουαρέκ και των Ισλαμιστών. Και στη, στη Μεθόριο με το Μαλί. Και εκεί ε, πραγματικά όχι μόνο η Λιβύη αλλά και η ευρύτερη περιοχή και η Αλγερία και άλλα κράτη της Βορειοφικής πραγματικά ε, πλέον ανθρωποιούνται. Και σε ό,τι αφορά τους αλαφιστές επίσης ίσως να εμπνευστούν από αυτά που έγιναν ε, στην ε, Αίγυπτο, αλλά και οι Βέρβεροι και αυτοί κάπως απομονώνονται και ίσως και αυτοί εξαγερδούν. Τώρα, ο φεντεραλισμός από πολιτικής πλευράς ε, ίσως είναι κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει να καταλαγιάσουν κάπως ε, όλες αυτές ε, οι από παλαιοτά των ετών ε, διαφορές. Αλζανούση ε, φαίνεται ότι θέλει να βοηθήσει τη χώρα του. Δεν ξέρω μήπως και οι βασιλείς θα μπορούσαν ενδεχομένως να επιστρέψουν για να μπορούν να διαδραματίσουν ένα ή μη ε, με έναν ρόλο μεταβατικό ή κάπως, όπως έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Και τι γίνεται με την οικονομία. Πρέπει να ξεκινήσει ε, πάλι η παραγωγή πετρελαίου. Ίσως χρειάζονται και διεθνή χρηματοοικονομική βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα ένα ερώτημα στον κύριο Λάμπστορφ σε πολλές νέες δημοκρατίες, αναδυόμενες δημοκρατίες, ομάδες προβληματισμού ή ιδρύματα από τη Δυτική Ευρώπη και από τις ΗΠΑ ε, έχουν δραματίσει ένα σημαντικό ρόλο. Ένα παράδειγμα είναι η Αίγυπτος, όπου υπήρχαν διάφορα προβλήματα και δεν ήταν καθόλου ξεκάθαρη ποια ήταν η θέση και το έργο αυτών των ε, δεξαμενών σκέψης και διαφόρων ιδρυμάτων. Τι πιστεύουν τα βασικά πολιτικά κινήματα για τέτοιου είδους ε, ιδρύματα ή think tanks που υποτίθεται ότι εργάζονται για τη δημοκρατία, για την εκπαίδευση τι γνωρίζεις για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας. Ξέρουμε ότι Κατάρ και Σαουδική Αραβία έχουν, κάνει μεγάλη, έχουν δώσει μεγάλη δημοσιότητα στην ε, χρηματοδότηση της ε, προεκλογικής εκστρατείας στην Αίγυπτο. Είναι γνωστό επίσης ότι αναμειγνύονται στις χρηματοδοτήσεις ορισμένων τμήματων της Συριανής αντιπολίτευσης της Συριακής μάλλον αντιπολίτευσης γνωρίζεις αν ε, αναμειγνύονται και στη Λιβύη. Απάντηση του κ. Ράμστορφ. Ευχαριστώ για την ερώτηση, ευχαριστώ και για το μεγάλο ενδιαφέρον που επέδειξαν οι συνάδελφοι. Ας αρχίσω με την ερώτηση για άλλες αποστολές που έχει σχέση και με τα think tank και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην χώρα θα γίνει και μια αποστολή από το κέντρο Κάρτερ, επίσης από το Έλλης που είναι Βρετανικό. Υπάρχει και ισχυρή παρουσία του National Democratic Institute ήδη από πολλών μηνών και έχουν συνεργασία με εγχώριες οργανώσεις παρατηρητών και συνεργασία με πολιτικά κόμματα. Δεν έχουν όμως επιτόπου ομάδες αξιολογήσεως, γιατί έχουν πάει εκεί να κάνουν άλλα πράγματα, αλλά συνεργάζονται με τοπικούς παράγοντες παρατηρήσεως. Αναμένω και τον Αραβικό Σύνδεσμο να εμφανιστεί λίγο πριν από την ημέρα των εκλογών και εμείς θα συνεργαστούμε όπως κατά παράδοση το πράττουμε με τις αποστολές αυτές θα τους αναπτύξουμε το τι έχουμε μάθει έτσι ώστε να έχουμε δυνατότητα να αξιολογήσουμε στέρεα την ε, κατάσταση και να μπορούμε να βασιζόμαστε και σε πηγές όλων των αποστολών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι όλες αυτές οι αποστολές θα είναι σχετικά περιορισμένες με το ολιγάρισμο προσωπικό που διαθέτουμε δεν μπορούμε να είμαστε παντού. Εγώ πέρασα μόλις λίγες μέρες εκεί και επέστρεψα το Σάββατο το βράδυ. Γι' αυτό και είπα ότι οι παρατηρήσεις που έκανα ήταν μια προκατακτική εκτίμηση για το πώς θα προχωρήσει η εκλογική διαδικασία. Πρόκειται για μια χώρα η οποία βγαίνει από έναν εφιάλτη πολλών δεκαετιών σε ό,τι αφορά τις πολιτικές της δομές. Αν θα πρέπει να είναι κανείς αισιόδοξο ή απεσιόδοξο, εγώ προέρχομαι από μια ε, περιφέρεια στη Γερμανία που είναι γνωστό ότι είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Τώρα, για τους τα μέλη βασιλικής, της βασιλικής οικογένειας. Οι συνομιλητές μου δεν τους έχουν αναφέρει. Κάποια συζήτηση γίνεται σχετικά με τον ενδεχόμενο να επιστρέψουν. Ίσως κάποιοι να το σκέφτονται αυτό, αλλά εγώ δεν έχω δει να παίζει κάποιο ρόλο στην πολιτική συζήτηση. Τώρα για την τιμή του πετρελαίου, ναι, είναι γύρω στα 90 δολάρια βέβαια αυτή τη στιγμή. Η χώρα έχει αρκετά από θέματα που μπορούν να την στηρίξουν έστω και αν το βαρέλι παίζει τα 70-80 δολάρια. Αυτό που τους ενδιαφέρει πολύ είναι επικοδομητική στήριξη που να σέβεται τα κεκτημένα της Λιβύης ότι πρόκειται για διαδικασία η οποία ανήκει στη Λιβύη το πέρασμα αυτό από τον εφιάλτη σε μια δημοκρατική ζωή. Πάντως δεν νομίζω το, ότι το χρήμα θα είναι ε, πρόβλημα. Τώρα σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις προς ορισμένες ομάδες από άλλες χώρες υπάρχουν φήμες. Η αποστολή δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει μέσα στις ε, ε, δύο εβδομάδες που βρίσκεται επιτόπου οποιαδήποτε από τις ε, φήμες αυτές. Πάντως η χρηματοδότηση της εκστρατείας μας απασχολεί. Θα γίνει έλεγχος και αυτό είναι σημαντικό και ενδιαφέρον θα, θα κληθούν όλα τα κόμματα να υποβάλουν τους λογαριασμούς τους σε ένα εποπτικό όργανο μετά τις εκλογές. Θα δούμε βέβαια πόσο αποτελεσματικό θα είναι το όργανο αυτό και πόσο αξιόπιστο. Για την ώρα πάντως δεν μπορώ να πω ότι εγώ μπορώ να επιβεβαιώσω οποιαδήποτε από τις φήμες αυτές. Τέλος. Α, για τη Σαρία και το Σύνταγμα μια στιγμή. Και την επιρροή των Ισλαμιστών. Να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα η, η, λιβική κοινωνία είναι παραδοσιακή, δεν είναι εξτρεμιστική, είναι παραδοσιακή Ισλαμική κοινωνία. Οι, άνθρωποι εκεί σέβονται τις παραδόσεις, υπάρχουν βέβαια διαφορετικές αποχρώσεις για το πόσο κοσμική με την έννοια του λαϊκού είναι ορισμένη, πόσο παραδοσιακά θρησκευτική είναι άλλοι, θρησκευόμενη δηλαδή. Αυτό είναι το θεμέλιο, αλλά πάνω σε όμοια θεμέλια μπορεί κανείς να χτίσει διαφορετικά σπίτια. Η ιδέα ερμηνεία που δίνουν στον Ισλαμικό νόμο οι διάφορες πλευρές είναι και αυτή ένα τμήμα αυτού του πολιτικού ανταγωνισμού για τον Τσάρλς. Ιδιαίτερα στον Νότο, όπως είπα υπάρχουν και όπλα, υπάρχει και απουσία ελέγχου στα σύνορα προς το Μαλί είναι ένα θέμα πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το ξύπνημα της Αλκάιδα την κατάσταση στο Βόρειο Μαλί θα πρέπει να συζητηθούν αυτά βέβαια μέσα σε ένα πολιτικό πλαίσιο και το τελευταίο ζήτημα που έχω πάλι έχει σχέση με κάτι που είπε ο Τσάρλς ορισμένες ομάδες του πληθυσμού που φοβούνται ότι θα μείνουν απ' έξω από τη νέα κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Και βέβαια είναι ενδιαφέρον ότι η Λιβύη εκλέγει ένα πολύ περίπλοκο σύστημα που είναι μείγμα πλειοψηφικού και αναλογικού. Υπάρχουν δηλαδή και κόμματα, αλλά υπάρχουν και μεμονωμένοι υποψήφοι. Σε ορισ... στι περισσότερε εκλογικέ περιφέρειες οι άνθρωποι θα ψηφίσουν δύο φορέ. Στη Γερμανία είχαμε το σύστημα αυτό 60 χρόνια. Και ακόμη οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει ποιο, που είναι, ε, ποιο είναι το πιο σημαντικό, πιο σημαντικό που θα βάλουν, ας πούμε. Λόγω της περιπλοκότητας του συστήματος, γιατί και αυτό δεν είναι και γενική ισχύω, ορισμένες περιφέρειες έχουν το αναλογικό, άλλες το πλειοψηφικό. Με το σύστημα αυτό, ορισμένες μειοψηφικές ομάδες έχουν ήδη εξασφαλισμένες τις έδρες ε, στο, ε, αντιπροσωπευτικό σώμα, στο κοινοβούλιο που θα εκλέξουν δηλαδή. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτή η σύνθεση του εν τέλει σε όλους τους σχηματισμούς αυτούς. Ευχαριστώ. Εγώ πάντως πιστεύω ότι πρέπει να διευκρινιστεί αυτό το θέμα της χρηματοδότησης και κατά πόσον αυτή προέρχεται από τρίτες χώρες. Νομίζω ότι είναι σκόπιμο να γίνει μια γενική συζήτηση Έχαμε και τον Πρωθυπουργό του Κατάρ εδώ, ο οποίος εξηγούσε πώς η χώρα του συνεισφέρει στην διατήρηση της ειρήνης και της ελευθερίας στον κόσμο. Νομίζω ότι ήταν ορισμένε ερωτήσεις που μπορούσαμε να του κάνουμε και σε αυτόν. Ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Τι άλλο μπορείς να μας πεις. Στα διάφορα, λέει ο κύριος Λάμστορφ, έχει εγκριθεί τώρα το κείμενο. Εγώ θα το βάλω βέβαια και γραπτό αυτό και θα το διαβάσω. Η εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου στο Board of Governors νομίζω ότι το επιτύχαμε αυτό. Με διασφάλιση εννέα εδρών υπέρ των Ευρωβουλευτών στο Διοικητικό Συμβουλίο. Δεν είναι δηλαδή καθαρά θεσμική εκπροσώπηση, θα είναι και πολιτική. Γιατί πρόκειται είναι και ένα όργανο που έχει σχέση με τη διασφάλιση δημοκρατία. Σε παρακαλώ, Έλμπαρ, να θέσει το θέμα αυτό και στου προέδρου των πολιτικών ομάδων για να δει πώ θα γίνουν οι διορισμοί των μελών. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο Μπροκ. Η πρότασή μου θα είναι, αν έχουμε νέα μέλη, να ζητήσουμε από την διάσκεψη των προέδρων πολιτικών ομάδων να κατανείμουν νέα αυτές έδρες σύστημα, το σύστημα hunt στις πολιτικές ομάδες. Αυτός νομίζω είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος. Συμφωνείτε? Η ε, κυρία Γκόμης. Συμφωνώ με την πρότασή σας, απλά θα ήθελα να τονίσω όπως είπε ο Αλεξάνδερ το ρόλο που έχουν οι NTS από το Σεπτέμβριο στην Λιβύη πολιτικά κόμματα, κοινωνία των πολιτών και για την ε, εκλογική επιτροπή, την εφορευτική επιτροπή. Όλα αυτά είναι ε, δείγματα του τι μπορεί να πετύχει ε, το ΙΝΤΙΑ, δηλαδή αυτό το Ίδρυμα για τη Δημοκρατία. Γιατί είναι εκεί, είναι εκεί γιατί τους επιτρέπει ε, με, πολύ την πολύ ευέλικτη δομή που έχουν να κινούνται και να οργανώνουν. Είπατε κύριε Πρόεδρε ότι έχουμε εννέα έδρες. Νομίζω ότι οι δύο πηγαίνουν ε, εξοφίκιο ε, στον, στους πρόεδρους των Επιτροπών Ντρουά και Ντέβε. Άρα και για τις εννέα θέσεις ισχύει ο κανονικός ε, των ΤΕΟΝ ή μόνο για τις ε, επτά θέσεις. Γιατί αν είναι το δεύτερο, ε, οι πράσινοι μπορεί να έχουν δύο και εμείς να μην έχουμε καμία θέση. Αν εφαρμόσετε το κριτήριο ΤΕΟΝ θα ήθελα να ισχύει για όλους και για τους εννέα και όχι μόνο για τους επτά. Ο πρόεδρος δεν νομίζω ότι είναι οι πράσινοι, κυρίες θα πάρουν. Λοιπόν, εγώ θα επαναλάβω και οι εννέα θέσεις θα κρεθούν με, με βάση τον τεό. Τώρα αν κάποιοι θα πρέπει να είναι εξωφίκιο, θα πρέπει να βρεθεί ένα συμβιβασμός. Τι είχαμε κάνει με μια ομάδα εργασίας πρόσφατα θα το δούμε. Θα πρέπει να προέρχονται από τις ομάδες αυτοί που θα οριστούν εξοφίκιο. Let's Ας δούμε πώς θα το κάνουμε. Έχουμε εμπειρία. Επόμενη συνεδρίαση. Αύριο Αυτό που σας είχα πει δηλαδή. Θα μπορούσαμε να συνεδριάσουμε σήμερα, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε την ενημέρωση για το άτυπο συμβούλιο. Θα έρθει ο Δανός όμως Υπουργός αύριο στις 12 για να μας ενημερώσει για μία ώρα για τα αποτελέσματα. Που τότε θα έχουν ολοκληρωθεί. Εγώ σας εύχομαι καλή ημέρα και εγώ είχα μια πολύ καλή μέρα αφού έγινα για τέταρτη φορά παππούς.